Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι. Δεύτερη σύνοδος. Τραπεζική Ένωση, Κεφαλαϊκή Ένωση, ενιαία αγορά για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ε, θέλω τώρα να καλωσορίσω τον Νούκο Μπάση από το τμήματάκι στη DG Φίνσε, κύριο Μάρια, από την ΕΜΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ο κύριος Πάτσα, Μπούχαρτ Πάλτσε που είναι ο συντάκτης μας ε, της έκθεσης ε, ιδίας ε, πρωτοβουλίας για τα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Μας έδειξε ξεκάθαρα η οικονομική κρίση ότι είναι αδύναμο το ρυθμιστικό μας πλαίσιο και ότι σε, και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι είναι ατελής ε, η ολοκλήρωση οπότε οι στόχοι που έχουμε Τα μέτρα που παίρνουμε φυσικά τροποποιούν ε, τον τρόπο λειτουργίας ε, της εσωτερικής ε, αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το επίπεδο αυτών των αλλαγών και το πόσο φιλόδοξο είναι το θεματολόγιο μας για την Τραπεζική Ένωση, Κεφαλαϊκή Ένωση και την Ενιαία Αγορά απαιτεί να κάνουμε σαφή διάκριση αφενός ε, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πέραν αυτού απαιτεί και ε, στενή συνεργασία ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και τα εθνικά κοινοβούλια. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι καλό να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτή την συνεργασία και ως προς την νομοθεσία αλλά και ως προς ε, τον ε, πολιτικό και ε, οικονομικό έλεγχο. Αρχίζω με την Τραπεζική Ένωση. Είναι φυσικά το πλέον φιλόδοξο σχέδιο που έχουμε. Και ήταν οι βαθύτερες και ριζοσπαστικότερες αλλαγές που επιτύχαμε μέχρι στιγμής. Έχει νομοθετικό ρόλο το Κοινοβούλιο αλλά και σημαντικότατο ρόλο για το πολιτικό έλεγχο. Έχουμε τη διοργανική συμφωνία με την ΕΚΤ. Και θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε διαρθρωμένη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη εποπτεία μέσω των ε, ρυθμιστικών αρχών που έχουμε στον τομέα αυτό. Τρεις ε, είναι οι τομείς όπου τρία είναι τα ζητήματα για τα οποία ε, χρειάζεται εντατικότερη συζήτηση. Πρώτα τραπεζική ένωση και μετά κεφαλαιακή κτλ. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι θεμητή όρια ανταγωνισμού και πώς θα συμφιλιώσουμε την ανάγκη για, για προσέγγιση των εποπτικών πρακτικών, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε έναν υγιή πλουραλισμό, αν θέλετε, των ε, τραπεζικών μοντέλων στην Ευρώπη, με μεγάλες τράπεζες, μικρές τράπεζες, Ε, ο κίνδυνος, ο κίνδυνος των αγορών, των, ε, δανειακών προϊόντων. Δεύτερον, σταθερότητα και ανάπτυξη. Πώς θα βρούμε την ε, ισορροπία για να αποφύγουμε την προκυκλικότητα και τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία διατηρώντας την ανάπτυξη. Νομίζω ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση η Επιτροπή κατέθεσε νέο πακέτο για την ε, τροποποίηση ε, για τα ίδια κεφάλαια. Υπάρχουν και διατάξεις ε, φιλοαναπτυξιακές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση μικροδομών και πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά με τις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις ε, της Βασιλείας, γιατί και θα είναι απόσπαστο κομμάτι της ε, διαδικασίας. Χρειαζόμαστε ένα, ε, ε, μια ισορροπία γιατί υπάρχει αυτή η πτυτικότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και ταυτόχρονα, όπως είπαμε και στο ψήφισμα της Ολομέλης, χρειαζόμαστε ισορροπία, ώστε ε, με τη ρύθμιση να μην πνίξουμε τα διαφορετικά τραπεζικά μοντέλα που υπάρχουν, υπάρχουν στην Ευρώπη. Τρίτον, περίπλοκα ζητήματα όπως η MPL ε, για την ε, εκαθάριση των τραπεζών. Οι κανόνες μας επιτρέπουν ένα ε, περιθώριο ελιγμών, αλλά τι μπορούμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, ε, μεταφοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κόκκινων δανείων. ε, διαβάζουμε τα σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε ποια είναι η δική σας άποψη. Κάποιες διευκρινήσεις δηλαδή. Μπορούμε να έχουμε εταιρείε διαχείρισης ε, στοιχείων ενεργητικού που ε, αυτά τα multi-purpose loans ε, θα, ε, θα προσδιορίζουν δηλαδή την αγοραία αξία αυτών των δανείων και πώς θα προσεγγίζουν αυτά τα προϊόντα συνέχεια οι τράπεζες. Αυτός ο μηχανισμός πώς θα λειτουργήσει για τον προσδιορισμό της τιμής. Ε, κρατικές προμήθειες, σχετικοί κανόνες, εξάντε, εξπόστ, προσδιορισμός των κοινών πόρων. Πολύ σημαντικά ζητήματα όλα αυτά και ελπίζω να μπορέσετε εσείς να μας πείτε κάτι διευκρινιστικό. Τελικά στάδια της Τραπεζικής Ένωσης είναι το ε, επόμενο θέμα που θέλω να θίξω. Υπάρχει ασυμμετρία ανάμεσα στη, στους κοινούς κανόνες και τα κοινά θεσμικά όργανα αφενός και αφετέρου των εθνικών πόρων ανισορροπία ανάμεσα ε, στο περιορισμό του κινδύνου και τον επιμερισμό του κινδύνου. Επισημαίνεται πόσο σημαντικότερες πρέπει να είναι οι προσπάθειες ε, για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο, να διαρρήξουμε αυτό το, αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο εθνικό χρέος και το χρέος των τραπεζών. Το backstop ε, το αποθεματικό που θα χρησιμοποιείτε, το έντις, ε, ο μηχανισμός εγγύησης των καταθέσεων. Επεξεργαζόμαστε την πρόταση για το έντις. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με σύνεση και ε, θα είναι ιδιαίτερα συζητήσεις μας ε, με τους εθνικούς βουλευτές κατόπιν ολοκλήρωση της Κεφαλαϊκής Ένωσης, ε, ολοκληρωμένες αγορές, ε, μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης. Αυτό θα είναι υποφελής για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, ε, δημιουργία αυτής της αγορές για όλα τα κρατημέρια είναι το επόμενο λογικό και σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Ε, φυσικά το κανόνας, ε, το εγχειρίδιο για την ενιαία αγορά ε, παραμένει προτεραιότητά μας. Έχουμε το σχέδιο δράσης που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς εγκρίναμε ε, στην Ολομέλεια. Ο κ. Ε, θα σας μιλήσει για την έκθεση πρωτοβουλίας μας ε, για θέλουμε να εντοπίσουμε τα κενά και τα παραθυράκια που μπορεί να υπάρχουν και στι αρνητικές επιπτώσεις σχέση με το βάρος απόδειξης. Το Νοέμβρη δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρόταση για το βάρος των αποδείξεων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, και έδωσε κάποιες απαντήσεις σε σχέση με αυτά που αναφέραμε εμείς ε, στο ψήφισμά μας ε, και πολλά επιμέρους στοιχεία του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστούν καλές απαντήσεις για την Κεφαλαϊκή Ένωση εξεργάζεται διάφορα νομοθετήματα για να τα προτείνει Έχουμε ήδη αρχίσει τις ε, διαπραγματεύσεις ε, στα πλαίσια τριμερών ε, διαλόγων για την τιτλοποίηση παραδείγματος χάρη και τα venture capitals, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και τα ομολογικά προϊόντα. Ο στόχος είναι να εντοπίσουμε τους, τα κενά που υπάρχουν στην ομοθεσία και η σένς που θα έχουμε για το CMU, για το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα, θα μας επιτρέψει να θέσουμε φιλόδοξους ε, στόχους. Θα είναι πλήρης η δέσμευση και η εμπλοκή μας στα επόμενα στάδια και θα έχουμε και άλλες δυνατότητες να τα συζητήσουμε αυτά με εθνικούς βουλευτές. Ο Γκομπάση θα πάρει πρώτος το λόγο, Ρία και μετά Μπούχορτ Μπάλτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ αγαπητοί και αυροβουλευτές. Με την πρόσκλησή σας μου δίνετε την ευκαιρία να σας αναπτύξω κάποιες σκέψεις για τα θέματα τα οποία ήδη σας παρουσίασε ο κύριος ε, Γκουαλτιέρης. Συγκεκριμένα πω γίνεται με την ε, ιδέα της ε, Ένωσης των Κεφαλαίων και να σας πω επίσης τι είναι με το Call of Evidence της Επιτροπής. Να σας πω πρώτα πρώτα τι γίνεται με αυτή τη σκανδάλη που ανέφερε ο κύριος Γκουαλτιέρη. Έχουμε ένα ψήφισμα της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπό την αιγύδα του κυρίου Μπάλτς πριν από ένα χρόνο υπήρξε το σχετικό ψήφισμα, αυτό το οποίο εγκρίνεται και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το πολύ σημαντικό ζήτημα του να διαπιστωθεί δηλαδή κατά πόσον το χρηματοπιστωτικό πλαίσιο όπως προέκυπτε από την ε, Ευρύτερη μεταρρύθμιση που έγινε κατά την ε, κρίση. Εάν αυτό, επομένως, το πλαίσιο ακόμη είναι δόκιμο και λειτουργικό. Αν επομένως για τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες τώρα βοηθάτε η χρηματοδότηση της ε, πραγματικής οικονομίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα αυτό είναι η αφετηρία μας και όσον αφορά αυτό το call for evidence είπαμε ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαβούλευση. Να σας πω κάποιες ιδέες μου. But already, since the beginning... Πάντως, έτσι για αλλιώς, από την αρχή της διαδρομής της Επιτροπής ε, ε, Juncker ε, δόχη μεγάλη προσοχή στην υπόθεση της Ένωσης των Χρηματοπιστωτικών Αγορών. Ήταν από τις κορυφαίες προτεραιότητες του πρόεδρου Juncker ακόμα και πριν τον ορισμό των επιτρόπων. Ακριβώ για να υπάρξει μία πιο ολοκληρωμένη αγορά για τις κεφαλαίες αγορές ούτως ώστε να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία όπου περισσεύει κεφάλαιο να πάει εκεί όπου λείπει. Άρα ο στόχος πάντοτε ήταν το πώς θα υπάρξει χρηματοδότηση πώ θα υπάρξουν ροέ προ την πραγματική οικονομία. Οπότε και εμεί ευθύ εξ αρχή αρχίσαμε να εντοπίζουμε κάποιε πρωτοβουλίε. Όποιε θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτευχή του στόχου. Πρώτα-πρώτα είχαμε ένα πρόγραμμα δράση το οποίο ξεκίνησε το 2015. Τότε εξαγγείλαμε μια σειρά πρωτοβουλειών μεταξύ των οποίων και την ανθεώρηση της οδηγίας για τα προσπέκτους αλλά επίσης ε, για το securitization ε, τιτλοποίηση, το, το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, του σχετικού κανόνε επομένω για όλα αυτά, ούτω ώστε να είναι όλα πιο αποτελεσματικά. Όλα αυτά επομένω δρομολογήθηκαν, όπω τα είπε και ο κύριο ε, Γκουαλτιέρη. Και τώρα έχουμε και επιπλέον πρωτοβουλίε πάντα αυτές αυτό το προγραμμα δραση δράσης. Οπότε βήμα-βήμα όλα αυτά τα υλοποιούμε. Το Σεπτέμβριο του 2016 επομένως ο έδινε σε κάποια ανακοίνωση όσον αφορά την ιδέα αυτή για την ένωση των αγορών και αυτό το κάνουμε για να ανταποκριθούμε στο ε, πρόβλημα το οποίο ε, εκκρεμούσε δηλαδή το κατά πόσον ε, έχει νόημα να υπάρξει αυτή η ένωση των κεφαλαίων αγορών μετά το δημοψήφισμα το αγγλικό και το Brexit φαντάζομαι στον ορίζοντα. Όμως είπαμε ότι χωρίς καμία επιφύλαξη η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, χρειάζεται αυτό. Και όχι μόνο χρειάζεται, αλλά θα πρέπει και να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει. Όπως επίσης θα πρέπει να βάλουμε τον πύχη των φιλοδοξιών μας ακόμα ψηλότερα για την υπόθεση αυτή της Ένωσης των Αγορών. Τώρα, το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ότι μελετήσαμε τις περαιτέρω πρωτοβουλίες, πέντε εξ αυτών και επίσης ε, μπήκαμε σε κάποια χωράφια που ήταν ταμπού μέχρι τώρα. Για παράδειγμα κάναμε κάποιες προτάσεις για να εναρμονιστούν κάποιες συγκεκριμένες πτυχές των εθνικών πτωχευτικών δικαίων. Και έτσι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιο καλόπιστο επιχειρηματία. Και αυτή μας η πρόταση τον Οκτώβριο πέρσι εγκρίθηκε. Επίσης τώρα μελετάτε το τι μπορούμε να κάνουμε για κάποιο είδου συνταξιδοτικό προϊόν πανευρωπαϊκό το οποίο θα έρθει να συμπληρώσει επικουρικά τα εθνικά συνταξιδοτικά συστήματα και ε, αυτό θα ήταν και επενδυτικό εργαλείο αξιόλογο στο μέλλον. Και αυτή η πρόταση ενδεχομένω ε, κατά το εναιστώσια του να εγκριθεί. Τα είπε και ο κύριο ε, Γκολτιέρη τώρα το αυτό το οποίο κάνουμε είναι προσπαθούμε να λάβουμε τα τελευταία στοιχεία από όλου του εμπλεκόμενου από όλου δηλαδή, όσου ενδιαφέρονται για αυτή την προβληματική. Είπαμε ότι έχουμε διαβούλευση ανοιχτή που ξεκίνησε πριν από κάποιε εβδομάδε και θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο του 2017. Όλα αυτά μπορείτε να βρείτε online στο website της διεύθυνσής μας. Και το θέμα είναι απλό. Γίνεται καταγραφή του τι ισχύει μέχρι σήμερα και προσπαθούμε να δούμε αν αρκούν αυτά που προτείνουμε και ή, ή αν χρειάζεται περαιτέρω πρωτοβουλία να αναλυφθεί. Πάντως, είναι σημαντικό το ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση τη μεσοπρόθεσμη του Ιουνίου ε, φέτος οπότε και έτσι ενδεχομένως ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την υπόλοιπη ε, περίοδο, για την υπόλοιπη θητεία αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορεί να φτάσει και ακόμα παραπέρα. Άρα ήρθε η ώρα οπότε οποιαδήποτε ιδέα, οποιαδήποτε πρόταση είναι καλοδεχούμενη. Θα πρέπει όλοι ε, να βοηθήσουν. Είπαμε ότι έχουμε εδώ πέρα μια εργαλειοθήκη, έχουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες, μη νομοθετικές πρωτοβουλίες και επίσης κάποιες πρωτοβουλίες που αφορούν ε, τη βιομηχανία, αφορούν ε, τα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάτι για όλους και όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν για αυτή την υπόθεση. Γιατί είναι κάτι που θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Άρα χρειαζόμαστε χείρα βοηθείας από όλους. Παράλληλα με όλα αυτά όπως σας είπα Έχουμε αυτή την ευρύτατη διαβούλευση για να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου. Έχουμε λάβει ήδη εκατοντάδες απαντήσεων στο σχετικό μας ερωτηματολόγιο και το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μπορεί να καταλάβει καλύτερα για το τι γίνεται, πώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, θα έχουν κάποιες επιπτώσεις και κυρίως αν έχουν αρνητικές. Ιδίως όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία ε, του κλάδου του χρηματοπιστωτικού και τα θετικά και τα αρνητικά και για την απασχόληση και για το θέμα του κατά πόσο όλα αυτά φέρνουν μια σταθερότητα στο σύστημα. Σας παραπέμπω μένω στην ανακοίνωσή μας του Νοεμβρίου. Δεν θα κάτσω τώρα να σας πω μία-μία τις πρωτοβουλίες που πρώτη θέμεθα να αναλάβουμε στη συνέχεια της, ε, της διαβούλευσης αυτής. Αλλά, αλλά να σας πω τους τέσσερις βασικούς τομείς όπου είδαμε ότι ενδιαφέρουν τους τέσσερις βασικούς στόχους που θα χαρακτηρίζουν τη δουλειά μας, είπαμε δηλαδή ότι πρώτα-πρώτα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι κανόνες δεν θα είναι φραγμός στην ε, ροή της οικονομίας και των ε, κεφαλαίων ότι ε, αυτού του είδους οι στόχοι της επιμελίας θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και θα πρέπει να διαλέξουμε τις μεθόδους που είναι οι πιο φιλικοί προς την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, να βελτιώσουμε τους τρόπους χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Και ακριβώς πως κύριος Γκουαλτιέρη θέλουμε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις ΜΜΕ όλες ακόμα και σε αυτές και ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύρια ευρώ και επομένως ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με κάποια σχέδια υποδομής, τι γίνεται με το τι ε, επίση θα πρέπει να κάνουμε σε σχέση με το νομοθέτημα υπαριθμών 2 για την πτώχευση και άρα θα πρέπει να έχουμε επενδύσεις σε υποδομές μακρόπνοες ήδη έχουν ξεκινήσει αυτές. Και από αυτά να είναι χρηστικά από τις επιχειρήσεις. Επίσης, αναλογικότητα. Πολύ σημαντική να λάβουμε υπόψη τους υφέρποντες κινδύνους για τις επιχειρήσεις. Δεν θα έχουμε μία λύση για όλους. Πάντοτε το λέγαμε αυτό. Αλλά έχουμε εμπειρικά στοιχεία ε, τα οποία ανέδειξε η διαβούλευση. Ότι δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως ε, την αναλογικότητα και να κάτσουμε έτσι να αναθεωρήσουμε την ισχύουσα ε, νομοθεσία τώρα να καταργήσουμε τη γραφειοκρατία όλο το διοικητικό άχθος όπου είναι άχρηστο ας πούμε ε, εκεί που έχουμε τα θέματα διαφάνειας, από ανακοίνωσης, υποχρεώσεις ε, δημοσιοποίησης διαφόρων στοιχείων, γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε βέβαια ότι οι νομοθετικές ευρωπαϊκές αρχές έχουν ό,τι πληροφορίες χρειάζονται για να κάνουν δουλειά τους. Αλλά την άλλη μεριά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε κανός είδους επικαλύψεις στην νομοθεσία και όλα αυτά θα πρέπει να απαλληφθούν από την νομοθεσία και έτσι η ζωή των επιχειρήσεων να είναι πιο εύκολη χωρίς βέβαια να διαταράξουμε και να φέρουμε αστάθεια στο σύστημα. Επίσης αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, το ρυθμιστικό θα πρέπει να είναι συνεπές, να μην αφήσουμε παραθυράκια, να μην έχουμε αντιφάσεις και επικαλύψεις. Έτσι θα γίνει η αναθεώρηση της νομοθεσίας. Εδώ βάζω τελεία και όποιος θέλει μπορεί να μου υποβάλει ερωτήσεις. Thank you very much, uh, Now... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ugo, τώρα Αντρέρια, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστησή μου που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Να ξεκινήσω με μία παρατήρηση. Πριν από 15 μέρες ήμουν στο Hong Kong για ένα συνέδριο και εξεπλάγινα από το πόσο αρνητική είναι η αφήγηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χρηματαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου νομίζω έχει συνεισφέρει στο να ενισχύσει ακριβώς ε, αυτή, την αντίληψη κατακαιρματισμού των αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν δούμε τα γεγονότα, το ότι έχουμε κάνει τα τελευταία 6 χρόνια, πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πράγματι, είχαμε κατακαιρματισμό εντός ενιαίας αγοράς, αλλά έχουμε αναλάβει νομίζω δράση σε τρεις άξονες. Έχουμε ενιαίους ε, κανόνες ε, με ρυθμιστική ε, επαναρρύθμιση. Εφαρμόζουμε επίσης και τους κανόνες των G20 και τους κανόνες των Σαντέρμετα. Ε, έχουμε, θα έλεγα, κάποιες ε, θεσμικές ε, παρεμβάσεις με το ΕΣΜΑ, EBA και το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και βεβαίως έχουμε και παρεμβάσεις στους ισολογισμούς και ενισχύουμε βεβαίως την ε, θέση, την κεφαλαϊκή ε, διαφόρων ε, ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε βλέπουμε πως υπάρχει μια βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βεβαίω δεν ισχύει το ίδιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω. Οι παρεμβάσεις δηλαδή τις οποίες ε, κάνουμε. Νομίζω πως ε, έχουν ένα αποτέλεσμα όσον αφορά την αποκατάσταση της ολοκλήρωσης των χρηματαγόρων. Τώρα ως πρόεδρος Μεκτής Επιτροπής να πω πως ε, σημαντικό είναι ότι η μεικτή αυτή επιτροπή έχει και τις τρεις εποπτικές αρχές και το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και την Κομισιόν και κοιτάμε ζητήματα οριζόντιου ενδιαφέροντος και εστιάζουμε σε κοινή τακτική αξιολόγηση κινδύνου, πάρα πολλή δουλειά επίσης για την προστασία των καταναλωτών γίνεται από κοινού, επίσης και ζητήματα ρυθμιστικά κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν παραδείγματος χάρη την διπλοποίηση ή τις υποδομές των αγορών. Οπότε και η κοινή μας εργασία πήγαινε αρκετά καλά. Τώρα, στο χρόνο που μου απομένει, θα ήθελα να εστιάσω σε τρεις ε, τομείς. Πρώτα απ' όλα, τις ε, τράπεζες ε, και τις αγορές ε, στην Ένωση των Χρηματαγών και τις νέες τεχνολογίες επίσης και πώς θα επηρεάσουν και την ρύθμιση αλλά και τις δομές των χρηματαγορών. Να ξεκινήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα με τις τράπεζες. Από θεσμική σκοπιά η Τραπεζική Ένωση ως ένα βαθμό Ε, καθιστά ακόμη πιο σημαντικό αυτό το οποίο είπατε στην εισαγωγή σας κύριε Πρόεδρε γιατί η Τραπεζική Ένωση αυξάνει την ε, ζήτηση για μια εναρμόνιση στο ρυθμιστικό πλαίσιο υπάρχουν τώρα βεβαίω κάποιε κεντρικέ αρχέ οι οποίε έχουν πάρα πολλέ δυσκολίε για να εφαρμόσουν διαφορετικού κανόνε ανάλογα με το που δραστηριοποιείται ε, ή έχει έδρα η κάθε τράπεζα που είναι υπευθύνη του. Οπότε Υπάρχουν συνεχώς αιτήματα για εθνικές, ε, για εθνικές ευχέρειες ε, και από την πλευρά επίσης της διάσωσης, ε, ο μηχανισμός π.χ. των απαιτήσεων υπαγωγής κτλ. Και από την άλλη έχετε δίκιο ότι υπάρχει ένα ποικιλόμορφο οικοσύστημα στις αγορές μας και βεβαίως υπάρχει αυτή η όθηση για ένα ενιαίο πλαίσιο για όλους. Οπότε πρέπει η αναλογικότητα νομίζω να αποτελέσει ένα στοιχείο κλειδί. Θεωρώ κατά την απόψή μου θα πρέπει να πάμε προς ένα ενιαίο ε, ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο όμως θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ε, απαιτήσει, ε, στην πολυπλοκότητα, στον κίνδυνο που αποτελεί κάθε τράπεζα για το σύστημα, οπότε σκοπεύουμε να εκδώσουμε ως ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ένα έγγραφο διαβούλευσης προσεχώς. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω για τις τράπεζες, ε, το αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, Έχουμε κάνει πολλά όσον αφορά τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Νομίζω πως φέτος θα προσπαθήσουμε να δημοσιεύσουμε, θα έλεγα, το πρώτο σετ κανόνων. Έχουμε την πρωτογενή ε, νομοθεσία, τους δευτερογενούς κανόνες, τις κατευθυντήριες γραμμές της Τραπεζικής Αρχής και το πακέτο που είχε συμφωνηθεί ήδη από το 2009 Οπότε αυτή η δουλειά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Βεβαίως στην παρέμβαση στον τραπεζικό τομέα έχουμε τρία βασικά σκέλη. Πρώτα απ' όλα έχουμε κεφαλαιακή ενίσχυση. Δεύτερον να αναγνωρίσουμε ε, ποια είναι τα προβληματικά εκείνα στοιχεία. Και το τρίτο βεβαίως είναι να ξεκαθαρίσουν οι ισολογισμοί. Από αυτά τα τρία νομίζω τα δύο τα έχουμε κάνει. Έχουμε ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαϊκή επάρκεια, έχουμε αναγνωρίσει ποια είναι τα προβλήματα όσον αφορά τα στοιχεία των τραπεζών και υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα με την προσαρμογή. Οπότε υπάρχει βελτίωση, ο λόγος, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων πέφτει, αλλά είναι πολύ αργός ο ρυθμός βελτίωσης και αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα φτάσουμε τα επίπεδα προκρίσης μέχρι 8-9 χρόνια από σήμερα που είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και αυτό ήθελα ακριβώς να θέσω ακριβώς για την ισορροπία μεταξύ ρύθμισης και ανάπτυξης γιατί δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στο εάν οι κεφαλιακές απαιτήσεις ή άλλες απαιτήσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη. αλλά αυτό το οποίο πραγματικά εμποδίζει την ανάπτυξη είναι η αλλε απαιτησει εμποδιζουν την αναπτυξη αλλα αυτο το οποιο πραγματικα εμποδιζει την αναπτυξη ειναι η καθυστερηση στην προσαρμογή. Αν έχουμε τράπεζε οι οποίε έχουν φορτωμένου ισολογισμού με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν μπορούν να επιτελέσουν τη βασική του λειτουργία, να δανείζουν και να στηρίζουν την οικονομία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι εδώ πέρα. Έχουμε ήδη δημοσιεύσει την έκθεση που προτείνει τρει δράσει. Πρώτα απ' όλα να ενισχυθεί η ρυθμιστική πίεση και νομίζω πως ο Συμποπτικός μηχανισμός και η Κεντρική Τράπεζα ε, κάνουν πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα. Δεύτερον, το εθνικό νομικό πλαίσιο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να μην έχουμε μεγάλες ε, περιόδους αβεβαιότητας, ε, παραδείγματος χάρη για τις κατασχέσει π.χ. σπιτιών και βεβαίω να δούμε το ότι θα γίνει στη δευτερογενή αγορά. Δεν μπορούμε να πιέσουμε τι τράπεζε να πωλήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αν δεν υπάρχει αγορά για να γίνει κάτι τέτοιο. Και τώρα έχουμε μόνο λίγου εξειδικευμένου επενδυτέ που έχουν την γνώση και του πόρου να επενδύσουν σε αυτέ τι αγορέ γιατί δεν υπάρχουν επαρκεί πληροφορίε και η δομή να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε η πρότασή μα είναι ε, και η προσωπική μου άποψη και την ανέφερα ε, και στι παρατηρήσει μου στο Λουξεμβούργο είναι ότι αν δείτε όλε τι κρίσει στην ε, η Ιαπωνία, στη Σκανδιναβία δεκαετία του 90, στη ΣΥΠΑ, αλλά και στην Ιρλανδία, στην Ισπανία εντό τη Ένωση, όταν έχουμε πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια για τα οποία πρέπει να φύγουν, θα έλεγα, από του ολογισμού των τραπεζών, συνήθω οι εταιρείε διαχείριση τέτοιων στοιχείων ενεργητικού είναι οι μόνε οι οποίε μπορούν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία και πρέπει να δούμε πώ θα αναπτύξουμε ένα κοινό υπόδειγμα ή μια κοινή προσέγγιση για τέτοιες ε, εταιρείε και να προσπαθήσουμε να κινηθούμε προς τα εκεί. Τώρα, να περάσω στην Ένωση των Κεφαλαίων Ο Ούγκο τα είπε, δεν έχω να προσθέσω πολλά. Να πω ότι για εμάς είναι σαφές ότι η κρίση έδειξε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται πάρα πολύ από την χρηματοδότηση από τις τράπεζες και αν κολλήσει αυτός ο διάβλος υποφέρει η ευρωπαϊκή οικονομία οπότε πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί διάβλοι χρηματοδότησης των οικονομιών. Έχει μεγάλη σημασία επίσης και για να μοιραστεί ο κίνδυνος, να υπάρξει μια διασπορά κινδύνου, οπότε έχει ε, δίκιο εδώ πέρα η Κομισιόν ότι αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο για την νομισματική ένωση παρά για την ενιαία αγορά. Και εδώ πέρα έχουμε κάνει κάποια δουλειά για να στηρίξουμε την ε, Κομισιόν ε, και τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την τιτλοποίηση, για τα προσπέκτους, ε, για τον κανονισμό. Σχετικό, η ΕΟΠΑ επίσης έχει κάνει μια πρόταση για μια πανευρωπαϊκή αγορά συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια ολοκλήρωση της αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Τώρα για τις νέες τεχνολογίες. Βλέπουμε εδώ πέρα γρήγορες ε, τεχνολογικές αλλαγές και προκλήσεις και νέους παίκτες οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά και μικρές νέες εταιρείε εξειδικευμένες και γίγαντες ε, τεχνολογικούς γίγαντες ε, που δεν λειτουργούσαν παραδοσιακά στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτό καλό νέο σε ένα βαθμό γιατί βεβαίως θα ωφεληθούν οι καταναλωτές ε, των υπηρεσιών και όσον αφορά το κόστος και την πρόσβαση υπηρεσίες βεβαίως ε, τίθεται το ζήτημα για εμάς ε, τις ρυθμιστικές αρχές της προστασίας των καταναλωτών, της ασφάλειας των πληρωμών και να διατηρηθεί όπως θα έλεγα μια επαρκής περίμετρος ε, εποπτείας. Οπότε, όπως σας είπα, πέρσι είδαμε παραδείγματο χάρη την ε, αυτοματοποίηση στις ε, σύμβουλες, τα big data, το μεγάλο όγκο δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται και συλλέγονται από διάφορες πηγές όπως τα κοινωνικά μέσα και ορίζουμε επίσης το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει μια πρωτοβουλία για την χρηματοπιστωτική τεχνολογία. Θα μείνω σε αυτά βεβαίω. Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μεγάλε αλλαγέ και ζητήματα και για την δομή των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών και για την ε, τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα το παρακολουθήσουμε στενά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο στην Ολομέλεια εγκρίναμε το σχετικό ψήφισμα και ζητήσαμε ρύθμιση της αγοράς. Ήταν ευρία η πλειοψηφία, ο Γκομπάση και άλλοι χαιρέτησαν αυτή το ψήφισμα ως θετικό βήμα και ε, προέκυψε και αυτό το call of evidence όπως ονομάζεται. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα από την Ολομέλεια ε, σε επίπεδο Επιτροπής και Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών είναι δεδηλωμένοι οι στόχοι. Ε, περασμένα χρόνια ε, έχουν ελεγχθεί οι επιπτώσεις της κρίσης και κυρίως οι επιπτώσεις επί της πραγματικής ε, οικονομίας και βλέπουμε επίσης πώς επηρεάζεται ο ανταγωνισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και επίσης βλέπουμε κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια προσέγγιση που βασίζεται σε προσμέτρηση του κινδύνου. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών ε, Υποθέσεων προσπαθεί να συνδέσει τα διάφορα κομμάτια του παζλ της ε, νομοθεσίας ε, για τους επιμέρους αυτούς τομείς. Βλέπουμε μέτρα ρύθμισης. Ε, διαπιστώνουμε πού έχουμε εκπληρώσει τους στόχους μας και πού όχι. Προσπαθούμε να καταργήσουμε τις επικαλύψεις και επίσης προσπαθούμε να επιδιώξουμε ε, να μην έχουμε σκοτεινή και διαφανή νομοθεσία. Το ίδιο επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το θεματολόγιο Refit. Ε, ex post ε, ε, αποτιμούνται οι συνέπειες των νομοθετημάτων και επικεντρώνει την προσοχή της λοιπόν σε αυτή την απλούστευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να το επισημάνω απευθυνόμενος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτό το call of evidence από το Νοέμβρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι αναφέρθηκε ήδη αυτό, έχουμε ε, το ε, υπόβαθρο, αλλά λείπουν πολλά στοιχεία ε, και δεν μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν ιδιαίτερα φιδωλή σε σχέση με τα στοιχεία που μας έδωσε για να υποστηρίξει αυτήν την για τις νέες νομοθεσίες. Ε, ζητούμε μια ξεκάθαρη πρόταση για να μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε μεταξέλιξη της κεφαλαιακής ένωσης και να επιτύχουμε και τους, στόχους, ε, τους αρχικούς στόχους της Τραπεζικής Ένωσης. Θα βασιστούμε στην αξιολόγηση αντε και ex διότι μόνο έτσι θα εγγυηθούμε ότι οι προτάσεις για την σταθερότητα, για την προστασία των επενδυτών και για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών θα μπορέσουν να ευοδοθούν και ε, θα επιτύχουμε την ενιαία αγορά, η οποία όμως θα είναι ευνοϊκή για όλους τους παίκτες, ακόμη για τους παίκτες μικρού και μεσαίου μεγέθους. Ε, έχουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, οποία θα θέλουμε να επισημάνουμε μέσα στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Παραδείγματος χάρη ε, εξέταση της αρχής αναλογικότητας ε, συστηματικά μία φορά το χρόνο τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνεται αυτό και στην ανακοίνωσή τη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαλείται νομοθετήματα που θα έπρεπε να εξεταστούν από την οπτική γωνία της αναλογικότητα. Ε, σίγουρα, εφόσον είμαστε συνομοθέτες, ε, χρειαζόμαστε αυτές τις αξιολογίες για να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Ε, ζητήσαμε ένα ευρύτερο πλαίσιο λοιπόν για την εξέταση της αρχής αναλογικότητας και όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παίκτες small banking box, small insurance box ε, ή οποιαδήποτε άλλα μικρά πακέτα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζονται από αυτή την οπτική γωνία. Θα ήθελα λοιπόν και σήμερα να δράξω την ευκαιρία και να απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να χαράξει το δρόμο λοιπόν προς μεγαλύτερη αναλογικότητα. Τρίτο σημείο που είναι σημαντικό για μένα, στη, στο ψήφισμά μας ε, μιλήσαμε για ένα συνεπές ε, πλαίσιο, διότι για τις τρίτες χώρες έχουμε ένα... Ε, κατακαιρματισμένο τομείο, το οποίο και θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο για να στοιχειοθετήσουμε και τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις μας με ε, τρίτες χώρες. Ανάλογα με τον ε, το κλάδο, ανάλογα με τον τομέα ή και ανάλογα ε, με τις πολιτικές συνθήκες ε, διαφέρουν οι ρυθμίσεις. Ε, θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε επί αρχών που θα μπορέσουμε εξάντε να επαληθεύσουμε και έτσι θα δίνουμε μια εντύπωση μεγαλύτερης διαφάνειας και θα έχουμε δυνατό, μεγαλύτερη δυνατότητα διαμόρφωσης των μελλοντικών εξελίξεων γιατί μην ξεχνάμε και το Brexit τα επόμενα δύο-τρία χρόνια χρόνια θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουμε τα επόμενα χρόνια θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, ε, το συνδυάσουμε αυτό και με την, τις αρνητικές ενδεχομένως εξελίξεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε από πλευράς των ΙΠΑ. τέταρτον, αναφερόμαστε σε μια διαφανέστερη, καλύτερη νομοθετική διαδικασία. Και τώρα ε, δεν ε, ε, μιλάμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δίνει το στίγμα επειδή έχει την νομοθετική πρωτοβουλία και που φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την ρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Όχι, απευθυνόμαστε και σε ευρωπαϊκές αρχές που ε, έχουν κοινή με τους νομοθέτες αρμοδιότητα βάσει της νομοθεσίας. Ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε ιδιαίτερα έντονες συζητήσεις με τις ευρωπαϊκές αρχές και έχουμε αυτό το σκρούτινι σλόδο όπου ε, ε εξετάζουμε την εφαρμογή των νομοθεσιών με τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και με ε, τα πρότυπα, τα τεχνικά πρότυπα έχουμε θεσμοθετήσει πλέον την συνεργασία μας αλλά υπάρχει και η ελεύθερη εντολή όπως μπορώ να το εντοπίσω, όπως μπορώ να το ονομάσω που προβλέπεται για την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή επίσης ε, υπάρχουν πράγματα που ε, διαπραγματεύεστε αποκλειστικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, όμως, εάν δεν εγκληθούν εγκαίρως αυτές οι προτάσεις ε, και από το συνομοθέτη, το αποτέλεσμα θα είναι... Ε, ε, να μην εκπληρωθούν οι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οπτικής Αρχής. Με τους συναδέλφους σας, με τον κύριο Ενρία και τους υπόλοιπους συναδέλφους από την ΕΣΜΑ, είχαμε περιπτώσεις όπου διαφωνήσαμε, ε, αναγκαστήκαμε να διαφωνήσουμε. Ε, τέλος, για να μην υπερβώ και το χρόνο μου, ε, ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε μια ανταλλαγή με τους εθνικούς βουλευτές ε, και με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Χαιρόμαστε για αυτή την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων. Και ε, συνηθίζουμε να έχουμε έντονες συζητήσεις ε, και με την ΕΜΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και υπάρχουν ρυθμίσει διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές αρμοδιότητες και για να ολοκληρωθεί το παζλ με επιτυχία πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε επιτυχώς όλοι μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπάλτς. Τώρα αρχίζουμε με τους ομιλητές. Φαβιέν Γαλλία. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε, επιτρέψτε μου να επικεντρώσω την προσοχή μου στο θέμα των συνεπειών του Brexit. Κύριε Μπάση κύριε Ενρία, μας εξηγήσατε τι διακυβεύεται. Και εσείς ιδίως κύριε Ενρία μας ε, δώσετε μια εικόνα αυτής της κατάτμισης της ε, κεφαλαίου αγοράς που θα δοθεί προς τα έξω γιατί ο τομέας στη Βρετανία είπε πρόσφατα ότι δεν θέλει κάποιο είδους δικαιώματα διαβατηρίου για το σύνολο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και είπαν ότι θα επικεντρωθούν σε στοχευμένες δράσεις ανακλάδο και αναπροϊόν. Δεν θέλουν να έχουν ε, το καθεστώς να τους διέπει της τρίτης χώρας. Θέλουν δηλαδή συγκεκριμένη συγκρότηση. Και κατά τη γνώμη σας, ακριβώς τι χρειάζεται τώρα ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Ευρώπη τον 27 ή τον 28 με ή χωρίς την Βρετανία, ούτως ώστε να κρατήσει αυτήν την αξιοπιστία και σταθερότητα που έχει τι θα πρέπει να γίνει στις συνομιλίες με τους Βρετανούς ούτως ώστε να διασκεδαστούν οι ανησυχίες για τον ε, τομέα γιατί είπαμε ότι εφαρμοστεί ο θα είναι το Βρετανικό εν προκειμένου. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκουργέρη. Ε, σοσιαλδημοκράτης Ιταλός. Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ότι η εξέλιξη της ε, Χρηματοπιστωτικής Ένωσης είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα δημιουργήσει ε, συλλογικά κέρδη για την Ευρώπη. Ακόμη όμως δεν έχουμε φτάσει στην ολοκλήρωση αυτής της ε, ένωσης. Ακόμα στη είμαστε στην αρχή της διαδρομής. Οι καθυστερήσεις όμως αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Έτσι, αναδύονται κίνδυνοι. Ακόμα και για το ευρώ και την επιβίωσή του. Επομένω, χρειάζεται να αναλυθεί η δράση κατεπηγόντως. Και έχουν πολλές επιλογές σχετικά με αυτό. Για να δούμε για την Τραπεζική Ένωση που έχει υποθεί πολλές φορές ότι βρίσκεται στη μέση της διαδρομής. Δεν έχουμε κάποιο είδους ε, ε, δημοσιονομικό backstop για κάποιες κρίσεις, δεν υπάρχουν εγγύσεις επίσης για τις καταθέσεις ακόμα. Οπότε εδώ και μήνες γίνονται κάποιες προσπαθίες, αλλά όλες οι χώρες είναι εκτεθειμένες όσον αφορά κάποια καταιγίδα, κάποια κρίση αν συμβεί και πώς μόνη κάποια χώρα μπορεί να το κάνει. Είδατε τι έγινε το 2009-2010. Είχαμε πάρα πολλέ αρνητικέ συνέπειε. οπότε γι' αυτό σας λέω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η εξασφάλιση και εγγύηση των ε, καταθέσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί σαν νομοθετική πρόταση της Επιτροπής που υπάρχει. Να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Όμω, ακόμη πιο σημαντικό από αυτό είναι να υλοποιηθεί ο μηχανισμός, ο ενιαίος μηχανισμός της επίλυσης των διαφορών. Έτσι θα εξασφαλιστεί η διάσωση των τραπεζών που πάσχουν. Έτσι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και αν κανείς ανατρέξει στην τραπεζική ιστορία θα δει ότι είναι σαφές ότι σήμερα αυτού του είδους ο μηχανισμός της επίλυσης των διαφορών είναι ανεπαρκής και αν χτυπήσει και κάποια τραπεζική κρίση πάλι θα είναι ανεπαρκής και γι' αυτό σας λέω μπορούμε κάπως να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε τον μηχανισμό και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε αυτού του είδους τη δημοσιονομική εξασφάλιση, τον backstop και να υπάρχει κάτι το οποίο να υποστηρίξει αυτό το Ταμείο Επίλυσης των Διαφορών. Και να είναι πιο ανθεκτική η Τραπεζική Ένωση. Αν επομένως συμφωνούμε και ε, τότε θα πρέπει να δούμε το πώς βέβαια και αυτή η προσπάθεια θα περιφέρεται από κάποιο είδους υποχρέωση δημοκρατικής ε, λογοδοσίας για απόδοση λογαριασμών. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω το πάνελ, τι σκέφτονται, πώς το βλέπουν. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια τέτοια λύση για αυτό το πρόβλημα. Μια που σήμερα στην Ευρωζώνη χρειάζεται να υπάρχει αυτού του είδους το fiscal backstop, αυτού του είδους η δημοσιονομική πλαίσιο για την ενδεχόμενη κρίση που μπορεί να χτυπήσει. Βέστρουντ, από τη Σουηδία. Σοσιαλδημοκράτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ε, να εξασφαλίσουμε ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων όπως και για τα πρόσωπα και για τα αγαθά. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν νομοθετική ρύθμιση και από πλευρά ε, Σουηδικού Κοινοβουλίου υποστηρίζουμε τις περισσότερες κινήσεις που γίνεται για την Τραπεζική Κεφαλαιακή Ένωση. Υπάρχει όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα πάντα ανακύπτει ε, σε σχέση με άλλους τομείς ε, δεν έχουμε κάνει αρκετές ε, προσπάθειες για την γραφειοκρατία. Παραδείγματο χάρη για την κεφαλαιακή ένωση και χρηματοπιστωτικές αγοράς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι θεσμικοί φορείς αλλά και μικρά, μικροί παίκτες που μπορούν να έχουν πολύ σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Είναι υπερβολικές οι ρυθμίσεις όμως και δεν τα καταφέρνουν με, αυτήν την, ε, με αυτό το γραφειοκρατικό άκτο. Ε, και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω τη σημασία την αρχή της αναλογικότητας ε, και επίσης να πούμε ότι γίνεται ιδιαίτερα επαχθή η διαδικασία κυρίως όταν εμπλέκονται και τα εθνικά κοινοβούλια. Λοιπόν, θα ήθελα να απευθύνω μια σχετική έκκληση και να πω ναι ότι αυτό το ορυφίτ και η καλύτερη νομοθεσία είναι κάτι που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια, αλλά θα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, ε, για την πραγματική οικονομία τελικά όταν ε, κάνουμε υπερβολικές ρυθμίσεις δυσχεραίνουμε περαιτέρω τη διαδικασία και την ε, καθημερινή ζωή αυτών των ε, μικρών παικτών. Ε, χρειαζόμαστε ένα σταθερό σύστημα επίσης για να έχουμε μια εύρυθμα λειτουργούσα κεφαλαιακή ένωση. Για τα, μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν μεγάλες δυσκολίες με αυτές τις περίπλοκες νομοθετικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μικέλ Βιέγκας, τώρα από την ΚΟΕ, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ. Ένα θέμα, μία ερώτηση που θέλω να απευθύνω γενικά στο πάνελ, όχι σε ένα συγκεκριμένο ομιλητή, σχετίζεται με κάτι που μας απασχολεί συνολικά. Ε, ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται αυτή η Τραπεζική Ένωση. Ποιος είναι ο στόχος. Ε, υποτίθεται ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τους ε, too big to fail, ε, τις υπερβολικά μεγάλες τράπεζες που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να πτωχεύσουν και ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα επιδεινώνοντας την, το λόγο ύπαρξης, αν θέλετε, της ίδιας της Τραπεζικής Γιατί τα λέω αυτά, διότι Τελικά ε, καρκινοβατούμε σε σχέση με μια τάση που προέκυψε μετά την ε, οικονομική κρίση, δηλαδή η ε, υπερρύθμιση του τομέα που τώρα υποχωρεί και δεν μιλάω εδώ για την προληπτική εποπτεία, δεν μιλάω για την ανάγκη ε, υπεράσπισης του τραπεζικού τομέα σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, αλλά μιλάω για τον πολλαπλασιασμό των χρηματοπιστωτικών προϊόντων μέσω της τιτλοποίησης που είναι και στη βάση ε, της οικονομικής κρίσης και τώρα επανέρχονται. Επανέρχονται αυτά τα προϊόντα ως ε, βασικό κομμάτι που θα μας βοηθήσει να τονώσουμε και πάλι τις επενδύσεις. Ε, λοιπόν, ε, αυτό θα πλήξει και πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως τώρα ρίχνουμε τα θεμέλια για μια μελλοντική ε, οικονομική κρίση ε, ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που γνωρίζαμε το 2008. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταϊκούρας, παρακαλώ, από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ουσιαστική, φιλόδοξη, όπως είπατε, παρέμβαση στην κατεύθυνση πρόληψης κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί χρηματοπιστωτική ένωση με βασικά συστατικά στοιχεία την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση των Κεφαλαγορών. Ήδη κατά την περίοδο της ελληνικής προεδρίας, το 2014, διαμορφώθηκαν δύο από τους πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτό που εκκρεμεί είναι ο τρίτος πυλώνας, με την υιοθέτηση και λειτουργία όμως ενός Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγύησης των Καταθέσεων αρχικά συμπληρωματικά με τα εθνικά συστήματα και μεταγενέστερα με έναν αμοιβοποιημένο μηχανισμό. Αυτός ο φορέας θα πρέπει να εδράζεται κυρίως στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 και όχι σε προτάσεις που συρρυκνώνουν τη ρευστότητα, ενισχύουν τη γραφειοκρατία, μειώνουν την αποτελεσματικότητα, μεταθέτουν χρονικά την επίλυση του προβλήματος, δεν αντιμετωπίζουν τα spillover effects. Παράλληλα, ταυτόχρονα, κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση μιας νέας δέσμης νομοθετικών προτάσεων με την ενσωμάτωση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών και προτύπων και τη διεύρυνση και ενδυνάμωση των πυλώνων της Βασιλείας με στόχο τη μείωση των κινδύνων. Σωστά όλοι αναφέρατε ότι κρίσιμο είναι να διασφαλιστεί η αρχή της αναλογικότητας. Ενώ οι ελάχιστε απαιτήσει για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμε υποχρεώσει πρέπει να διαμορφώνονται σε ρεαλιστικά επίπεδα, λαμβάνοντα υπόψη και την ανάγκη ορθολογική περίοδου προσαρμογή. Εξίσου όμω σημαντική είναι και η ψηφιακή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματο και η πρόταση για τη δημιουργία μια ένωση των κεφαλαιογορών με στόχο τη διεύρυνση και διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδίω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους που εμφανίζεται συρρήκνωση του τραπεζικού δανεισμού, κυρίως σε bank-based χώρες. Στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων θα μπορούσαν να εξεταστούν η αναθεώρηση και ο εξυγχρονισμός του πλαισίου προστασίας των επενδυτών στο πρότυπο του αντίστοιχου πλαισίου για τους καταθέτες και η ασφάλεια των συναλλαγών και η ανθεκτικότητα του συστήματος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. João Galamba, Portugal S&D. Ζωά Γκαλάμπα, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Πορτογαλία. Καλημέρα. Δύο ερωτήσεις έχω στον κύριο Ένερια της ΕΜΠΑ. Πρώτον, όπως είπε και ο κύριος Καλαιώτη τώρα, είμαστε σε αυτή την πορεία που δεν έχουμε κάνει τα απαραίτητα βήματα για να έχουμε την εγγύηση των καταθέσεων ακόμη, ε, ούτε και το fiscal backstop. Για να σημειωθεί πρόοδος Πρέπει να έχουμε επιπρόσθετες ε, κεφαλαιακές απαιτήσεις ε, για το δημόσιο χρέος από πλευράς δηλαδή των τραπεζών. Και αν το κάνουμε αυτό δεν θα επέλθει μεγαλύτερη αστάθεια διότι θα πούμε ότι ε, θα είναι ένα κομμάτι του ενεργητικού που τελικά θα χαρακτηρίζεται από κίνδυνο. Γιατί οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν αλλιώς σε επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ποιες λοιπόν θα είναι οι συνέπειες αυτών των ε, νέων μέτρων. Αν και αν χρειάζεται αύξηση του κεφαλαίου και όταν μιλάμε για διαχείριση του κινδύνου και ε, για διαχείριση του δημοσίου χρέους, ε, δεν θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκά ε, κριτήρια, διότι σε όλα τα φυσικά συστήματα και κυρίως αυτό που εντάσσεται σε μια οικονομική και νομισματική ένωση, θα πρέπει να λειτουργήσουμε χωρίς κίνδυνο. Αλλιώς δεν λειτουργεί το σύστημα, λοιπόν. Ποιο θα είναι αυτό το στοιχείο ενεργητικού χωρίς κίνδυνο που θα αντικαταστήσει το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, για τις bad banks και τα MPL, αυτά τα δανειά πολλαπλών χρήσεων. Επειδή είναι πολύ υψηλό ε, το κομμάτι των κόκκινων δανείων, τι θα γίνει, θα τα αγοράσετε σε fair value ε, και ε, θα μπορέσετε δηλαδή να καλύψετε τα κοινά που υπάρχουν. Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των MPL στην πραγματική οικονομία και ακριβώς πώς θα επηρεαστούν οι τράπεζες και γενικότερα ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας αν επιλέξουμε αυτή την άγουσα. Και κάτι άλλο. Έκανα μία πρόταση χθε. Δεν είναι δική μου η πρόταση, απλώς την μετέφερα χθε. Εξυγίανση των κοκκίνων δανείων στις ε, τράπεζες ε, μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες Δηλαδή, θέλω να πω αυτές οι προτάσεις που γίνονται για το πάγωμα των δανείων, πώ απλώ αναβάλουν το πρόβλημα. Ναι, σας ευχαριστούμε, λέει ο κύριο ε, Γκουαλτιέρη. Ε, ήδη έχουμε πάρα πολύ καλές ερωτήσεις, ε, οπότε θα πρότεινα να κάνουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων. Σας παρακαλώ όμω σύντομα, γιατί και πρέπει να τελειώσουμε στη μία και θέλουμε να κάνουμε και δεύτερο γύρο. Οι από τις ερωτήσεις για τον κύριο Ενρή, αλλά τέλος πάντων, ε, εγώ έχω να πω ότι η αναλογία αναφέρθηκε πολλές φορές. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι έτσι καλύπτουμε σφαιρικά τα πράγματα. 360 μοίρες για ασφαλιστές, για τράπεζες, για μάνατζες των περιουσιακών στοιχείων. Πολύ σημαντικό. Ναι, όλα αυτά επήγουν και η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει μια δυναμική περίπλοκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την νομοθεσία. Ξέρετε πώς είναι το σύστημα. Καμιά φορά παίρνει παραπάνω χρόνο από όσο θα θέλαμε. Για το Brexit τι να σας πω. Λέω απλώς ε, πιστεύω ότι είναι αδύνατο να προβλέψουμε που θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσει ακριβώ, αλλά από πλευρά Ένωση Κεφαλαίων θεωρούμε πω ε, εάν και όταν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τότε θα είναι ακόμα πιο σημαντικό οι 27 να έχουν την ε, Ένωση των Χρηματοπιστωτικών Αγορών. Και να υπάρχει μια τέτοια αγορά που να είναι ολοκληρωμένη και να καλύπτει και τους 27. Γι' αυτό σας είπα ότι εν ώψη του Brexit είναι ακόμα πιο σημαντική η Ένωση η χρηματοπιστωτική. Ο κύριος Ενρία. Πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνος. Να σας τα πω γίνεται πιο σύντομα. Όσον αφορά τις εταιρείες διαχείρισης ε, στοιχείων ενεργητικού, όπως ανέφερε ο τελευταίος ομιλητής, κοιτάξτε, τι ισχύει. Ε, βέβαια και η αξιολόγηση αυτών των ε, στοιχείων δεν είναι η αγοραία τους αξία. Αλλά αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για τις τράπεζες και για τους πελάτες τους. Και αν θεωρήσουμε ότι η πρόταση έχει ως στόχο το να έχουμε δευτερογενή αγορά αποτελεσματική και με αυτά τα στοιχεία ενεργητικού να μπορέσουμε να έχουμε αύριο καλύτερες τιμές. Άρα να υπάρχει κάποιο είδους γέφυρα, να πουλούν σήμερα οι τιμές σε κάποια αγορά αποτελεσματική και κάποια στιγμή να έχουμε ένα διάστημα τρία χρόνια όχι παραπάνω, οπότε αν είναι ψηλότερη η τιμή από την πώληση να αποζημιθούν οι τράπεζες ή όχι. Αυτά είναι κλασικές κινήσεις που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση για, τον, για την ανταγωνιστικότητα. Να μην αφαιρεθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα απομονωμένη η τράπεζα. Και επομένως... The current framework functioning, allowing Και άρα θα πρέπει να η ισχύση του προβλέπει οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια. Και να δούμε τι γίνεται και στις δευτερογενείς αγορές όσον αφορά τις πραγματικές τιμές το περιουσία των τραπεζών. Όσον αφορά την ολοκλήρωση τώρα της Τραπεζικής Ένωσης, όντως, συμφωνώ, υπάρχει πίεση, επίγει να ολοκληρωθεί το εγχείρημα, ό,τι εκκρεμεί και συζητείται τώρα αλλά να καταλάβουμε τι έχει γίνει, τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Πολύ σημαντικά έχουμε την αναγνώριση των προβλημάτων της περιουσίας, τα εποπτικά προβλήματα, ε, προσπάθεια να λειτουργήσει το σύστημα και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εποπτεία. Και όσον αφορά το πρόγραμμα για τις ε, εγγύησεις, μακροπρόθεσμα, έχουμε διαπιστώσει το παρελθόν ότι έχουμε την εκροή των καταθέσεων από κάποιες χώρες. Ε, αυτό δεν είναι καλό για το σύστημα συνολικά. Και ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε κάποια άλλα στοιχεία, άλλες μεταβλητές του συστήματος, που θα πρέπει να δούμε προς τα πού κατατείνουν. Γιατί δεν θέλουμε να καταλήξουμε στο σενάριο κατά το οποίο οι τράπεζες χρειάζονται χρήματα από τον δημόσιο κορβανά και το... θα πρέπει να είναι η εξαίρεση δηλαδή η ενεργοποίηση του συστήματος της ε, εγγύησης των καταθέσεων και να έχουμε διάσωση από τον ιδιωτικό τομέα όπως είδαμε πριν από μερικά χρόνια το Μπέιλιν δηλαδή τώρα συγγνώμη δεν κάψα κάποιες ερωτήσεις αλλά όσον αφορά το θέμα της περιπλοκότητας της νομοθεσίας σας επισημαίνω ότι δεκαετία του 90 ξεκίνησαμε με τη σύμβαση της Βασιλείας Παρθμονένου. Ήταν 40 σελίδες σύμβαση. Όμως άρχισαν τότε η παράκαμψη της νομοθεσίας και είχαμε τιτλοποιήσεις, ε, back-to-back ε, συναλλαγές ε, με διάφορους τρόπους. Κατεβλήθη προσπάθεια να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την πρακτική στις αγορές. Άρα γι' αυτό έγινε η νομοθεσία πιο περίπλοκη. Πολύ ωραία θα ήταν να πούμε ότι θέλουμε μόνο, υπάρχει μόνο το μετοχικό κεφάλαιο, μα όχι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολύ πιο σοφιστικέ και περίπλοκα εργαλεία. Ε, γι' αυτό και η νομοθεσία είναι αντίστοιχα περίπλοκη. Ακολουθεί και παρακολουθεί την εξέλιξη στην αγορά η νομοθεσία. Και ακριβώ όπω είπατε και οι περισσότεροι, γι' αυτό και χρειάζεται περισσότερη αναλογία και αναλογικότητα. Δηλαδή να νομοθετούμε αλλά να μην φορτώνουμε με υπερβολική νομοθέτηση της τράπεζας. Υπάρχει κάποιο είδους κανονισμό, κάποιο είδους κώδικας ψηφιακό που να ξέρουν οι τράπεζες τι ισχύει. και κάθε φορά να βλέπουν τι ισχύει. Βέβαια, μία μικρή τράπεζα θα πρέπει να συμμορφωθεί με 10% των διατάξεων ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε σχέση με μια μεγάλη τράπεζα. Εν κατακλείδη, όσον αφορά για το κατά πόσον τώρα έχουμε τάση για απορρίθμιση, κάτι που το ακούμε όλο ένα και περισσότερο και αλλού, συγκεκριμένα στη ΣΥΠΑ. Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, ότι έχουμε τέτοια τάση. Ας πούμε για την τετλοποίηση κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να έχουμε εύρυθμες αγορές, αγορές που να διακρίνονται από ασφάλεια. Τα στοιχεία ενεργητικού να είναι ξεκάθαρα και από κάθε άποψη να υπάρχει ασφάλεια στις αγορές. Μπάλτσα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σενεριά. Και εγώ δεν βλέπω μαύρα σύννεφα όπως είπε ο συνάδελφος ε, Πάτα από την, πάνω από την Ευρώπη όσον αφορά την απορρίθμιση. Αντιθέτως, δεν βλέπω να πηγαίνει το εκρεμές ε, προς την ε, άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι η απορρίθμιση, η προσέγγιση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές πως κάποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμείται κάτι τέτοιο, αλλά Κοιτάξτε, έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια με μεγάλη ένταση ε, στην Επιτροπή μας, ε, στο Κοινοβούλιο, προχωρήσαμε σε ρύθμιση των ε, χρηματαγορών και κοιτάμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα στην ε, πράξη. Αυτό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Κατόπιν για το θέμα της Ένωσης των Χρηματαγορών θέλω να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε ο Γκομπάση. Ε, κατά την απόψή μου πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο εγχείρημα και είναι σημαντικό και ούτως ή άλλως και ε, ειδικά δεδομένης της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και ξανατώνησε ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης πως ε, ως ε, Επίτροπος ε, για τις χρηματαγορές θέλει ακριβώς να ακολουθήσει την πορεία του προκατόχου του, του Λόρδου Χίλ και νομίζω πως είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα. Να προσθέσω ένα πράγμα. Σημαντικό για μένα. Η Ένωση των Κεφαλαγορών βεβαίως θα πρέπει να εξυπηρετεί την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω πως δεν πρέπει να επιτρέπεται να κάνουμε το λάθος να προωθήσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα αλλά αυτό το οποίο τελικά ε, έχουμε ως ισχυρά σημεία στην Ευρώπη να το αμφισβητήσουμε. Δηλαδή μια χρηματοδότηση η οποία θα γίνεται μέσω των χρηματαγορών δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπονομεύσει την παραδοσιακή θα έλεγα χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να έχουμε προβλήματα στην άλλη πλευρά γιατί είναι σαφές ότι και στην Ευρώπη ότι 70% της χρηματοδότησης προέρχεται από τις τράπεζες. Και νομίζω ότι θα πρέπει ακριβώς ε, να το έχουμε πάντα κατά νου αυτό. Τώρα για επιπρόσθετες απαιτήσεις, για επιπρόσθετες ε, κεφαλιακές απαιτήσει κάτι το οποίο έφερε ο συνάδελφο από την Πορτογαλία, πράγματι είναι ε, μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και η άποψή μου είναι η εξή ότι αυτό το οποίο θα γίνει στον επόμενο γύρο της ε, Βασιλείας, ε, στη Βασιλεία 4, πρέπει να μας απασχολήσει. Ε, υπάρχει μια βεβαιότητα αυτή τη στιγμή για το τι θα κάνει ο μεγάλος εταίρος την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είπα, και σήμερα δεν είμαι προσωπικά σε θέση να πω ότι θα πρέπει εμείς να επιβάλλουμε περαιτέρω κεφαλιακές ε, απαιτήσεις. Τελευταίο, Brexit. Πράγματι το ερώτημα της συναδέλφου Κέλλερ είναι θεμητό, δηλαδή Ποιο είναι, το ενδιαφέρον των αγορών. Πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά ακριβώς ε, το τι θα, ποιες αγορές θα παραμείνουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια θα είναι τα συμφέροντα μετά το Brexit, κάτι το οποίο θα πρέπει βεβαίως να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε και εμείς τα δικά μας τα συμφέροντα, δηλαδή στις ε, διαπραγματεύσεις το Λονδίνο θα παραμείνει οπωσδήποτε ε, ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο και μετά το Brexit, αυτό είναι σαφές, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απεμπολίσει τα δικά της συμφέροντα. Παραδείγματος χάρη να αναφέρω το ζήτημα του του clearing, ε, του euro clearing, δεν νομίζω παραδείγματος χάρη. Δύσκολα φαντάζομαι πως θα παραμείνει στην σημερινή του μορφή στο Λονδίνο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Έχουμε άλλους πέντε ομιλητές. Το πολύ δύο λεπτά παρακαλώ να μιλήσετε. Ραλφ Μπρινχάους, χριστιανοδημοκράτης από τη Γερμανία. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία ζητήματα. Πρώτο θέμα η ρύθμιση. Έχουμε εμείς αρκετές μεσαίου μεγέθους τράπεζες και θα πρέπει να υπάρχει η διπλή λεγόμενη αναλογικότητα, δηλαδή οι μικρές ε, τράπεζες ε, πράγματι να ε, υφίστανται και αυτές μια εποπτεία και να μην ασχολούμαστε συνέχεια μόνο με τις μεγάλες και πιο συστημικά επικίνδυνες τράπεζες χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι θα επιδοτούμε τις μεγαλύτερες με κάποιο τρόπο δεύτερον ασφάλιση καταθέσεων. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε κάποια στιγμή στον τρίτο πυλώνα. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει στη Γερμανία μεγάλη αντίσταση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και αυτό οφείλεται στο ότι δεν θεωρεί ο κόσμος ότι έχει προχωρήσει αρκετά ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας και υπάρχουν και κάποια ουσιαστικά προβλήματα. Ότι εξακολουθούν πολλοί ισολογισμοί τραπεζών να είναι φορτωμένοι με κρατικά ομόλογα και δεν έχουν επίσης κάποιον περιορισμό όσον αφορά τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν μέσω αυτών. Οπότε Υπάρχει ο κίνδυνο ότι χρησιμοποιείται αυτή η ιδίωδο για μια έμεση κρατική χρηματοδότηση. Επίσης και στη Γερμανία έχουμε πάρα πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια βάρη θα έλεγα του παρελθόντος και να προσπαθήσουμε να τα κοινωνικοποιήσουμε μέσω μιας ε, κοινή ασφάλισης είναι κάτι το οποίο βρίσκουμε οπωσδήποτε λανθασμένο και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχουν και εκείνες οι δομές ε, της διοίκησης η οποία σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το πρόβλημα το οποίο ανέφερα με τα κρατικά ομόλογα και να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Τέλος, εγώ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε κάποιο είδους ηθικό κίνδυνο, δηλαδή ότι δεν θα επιμετρούμε πλέον τον κίνδυνο όπως ε, θα έπρεπε γιατί θα υπάρχει πάντα η βαλβίδα εκτόνωσης η οποία λέγεται ακριβώς ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε θα πρέπει να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός. Γι' αυτό ακριβώς ε, είμαστε πολύ επικριτικοί Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Ο σας ευχαριστούμε. Ενρίκη Δίας ε, από την Πορτογαλία, Σοσιαλδημοκράτε. Γεια σα. Έχω τρει σύντομε ερωτήσει. Πρώτον, αυτή η κατάτμιση όσον αφορά το κρατικό χρέος. Πρώτα απ' όλα σε κλίμακα Ευρωζώνης και δεύτερον στην Ευρώπη γενικότερα. Έχουμε τώρα μια φάση μεγάλης πίεσης. Έχουμε αύξηση των ε, κεφαλαίων απαιτήσεων. Και λένε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ε, υγεία του τραπεζικού συστήματος. Όμως δεν έχουμε λύσει ακόμα τα διαφορετικά προβλήματα της ε, Τραπεζικής Ένωσης γιατί συνεχώς αναβάλουμε ε, τη θέσπιση του backstop και την εγγύηση των καταθέσεων. Οπότε αν μπορέσουμε αυτά τα κριτήρια να τα ενώσουμε, να τα συνενώσουμε. Ε, αυτό είναι κοινή ε, θέληση. Και να μην πληρώνουν την ύφη οι φορολογούμενοι. Να μην πληρώνουν αυτοί τη, τη, τη των τραπεζών. Αλλιώ όλε αυτέ τι προσπάθειε παραμένουν όνειρα θερινή νυχτό. Γιατί και στην Πορτογαλία. Το μάρμαρο το πλήρωσαν οι φορολογούμενοι και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και τις ενιαίες εποπτικές αρχές για να δώσουμε μία απάντηση. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξηθεί ο έλεγχος και τι μπορούμε να κάνουμε για να επιψευθεί η εφαρμογή των βασικών πυλών της Τραπεζικής Ένωσης. Πρώτον. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω το εξής η, αναθεώρηση της οδηγίας για τα ημεροπτικά φυλάδια. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνέταξαν μια θετική μεν έκθεση, αλλά τελικά περιορίστηκαν στο να διαπιστώσουν τις ελλείψεις όσο στην την εφαρμογή τη οδηγία για την ενημερωτικά φυλάδια. Ε, σε σχέση με την έκδοση χρέου και την αύξηση του κεφαλαίου υπάρχουν ακόμη πολλές ελλείψεις, κυρίως σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα, θα έπρεπε να έχουμε κάνει πολύ περισσότερα και ερωτώ το εξή. Μήπως χάνουμε μία ευκαιρία ε, να επαναδρομολογήσουμε αυτές τις κεφαλαιακές ε, ενώσεις ως εναλλακτική λύση στην ε, τραπεζική πίστη μέσα από αυτή την αναθεώρηση οδηγίας για τα ενημερωτικά φυλάδια. Ευχαριστούμε. Γεράσιμος Μπαλούρας, Ελλάδα, Αγκού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τραπεζική ένωση αλλά κάρτ δεν μπορεί να υπάρξει. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, εφόσον διαχέει το ρίσκο στον τραπεζικό τομέα και εγγυάται με τον ίδιο τρόπο τις καταθέσεις, σε όλα τα κράτη-μέλη σταθεροποιεί το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Είναι ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η υλοποίηση του τρίτου, τρίτου πυλώνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το EDIS θα πρέπει σταδιακά να έρθει σε πλήρες καθεστώς συνασφάλισης μέσα στα επόμενα 6 χρόνια, ώστε να είναι σε θέση να προστατευτούν οι μικροί και μεσαίοι καταθέτες. Τα τραπεζικά συστήματα, ακόμα και εκείνα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, πρέπει να γίνουν ασφαλή και με επαρκή ρευστότητα, ώστε να ανταπεξέλθουν σε μια ενδεχόμενη οικονομική συστημική κρίση. Έπειτα πρέπει να μην ξεχνάμε, συνάδελφοι, ότι αυτή η ανισομέρεια εγγύηση ανάμεσα σε διαφορετικά τραπεζικά συστήματα ανά την Ευρώπη προκαλεί μεταξύ άλλων και τη μεταφορά κεφαλαίων από τον Ευρωπαϊκό Νότο προς το πλεονασματικό και ασφαλή Βορρά. Γεγονός προκαλεί και έντονο πρόβλημα ρευστότητας. Αν οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς, τότε οι τράπεζες θέτοντας θέτοντά τους, εμείς δηλαδή εσείς, ένα πιο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα επανέλθουν στα παραδοσιακή τραπεζική και θα διοχετεύουν κεφάλαια, όπως είπε και ο πρόεδρο επενδύσεων ιδίω στι στις επιχειρήσει. επιχειρήσεις. Και τελειώνω με μια ερώτηση. Ποια είναι η αποψή σα για τι καθυστερήσει, στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος εγγύης καταθέσεων και στις προσπάθειες που γίνονται από συγκεκριμένα τραπεζικά συμφέροντα να το αποδυναμώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, David Coburn. David Coburn, Ευρωβουλευτής του EFTD. Ευχαριστώ κύριε Κουαλτιέρη. Άκουσα τον Σενιόρε Ενρία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που είπε ότι ε, στο Χονγκ Κόνγκ βλέπουν αρνητικά τις ευρωπαϊκές αγορές. Ε, δεν προξενεί εντύπωση, ειδικά μετά τον Brexit. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις υπερβολικές ρυθμίσεις της ε, ειλικρινά πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Έχετε σκεφτεί ποτέ το να μην παρεμβαίνετε σε επιχειρήσεις και να τις αφήσετε να λειτουργήσουν. Η υπερβολική ρύθμιση σκοτώνει τις αγορές. Αφήστε τα στις χώρες, στα κράτη. Γι' αυτό πηγαίνουν οι αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει μια ε, ελαφριά ρύθμιση. Και το Brexit θα επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Ο κεντρικός σχεδιασμός είναι επικίνδυνος, κύριε και κύριοι. Περιτέρω ολοκλήρωση σημαίνει περισσότερους κινδύνους. Αν υπάρχει μια κρίση, κάποιες τράπεζες σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικό μοντέλο μπορεί να επιζήσουν. Εάν είναι όλες συνδεδεμένες και παρόμοιες, όλες μαζί θα βουλιάξουν όπως όταν έσπασαν οι μπουλμέδες του Τιτανικού, ο οποίος ξέρετε, αν ε, ένας μπουλμές αν δεν είχε διαραγεί θα είχε παραμείνει στην επιφάνεια του Τιτανικού. Λοιπόν, γιατί πηγαίνουν οι αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Χονγκ Κονγκ, γιατί δεν υπάρχει υπερβολική ρύθμιση και συγκεντρωτισμός σαν την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα κινδυνεύει περισσότερο γιατί ο ένας τραβάει τον άλλον με την αλυσίδα και πέφτουν όλοι μαζί στον γκρεμό. Και κάνα δύο χώρες κινδυνεύουν να βγουν εκτός Ευρωζώνης και πρέπει να προετοιμαστείτε γι' αυτό και να σας ανισχύει περαιτέρω ολοκλήρωση. Η, Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία μου θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό το λόγο. Αλλά δεν θέμε να γειτονεύουμε με μια οικονομική καταστροφή δεν θέλουμε πραγματικά να υποφέρετε. Είναι μια καταστροφή θα είναι κακή και για μας. Προσπαθείτε λοιπόν, σας παρακαλώ, να αλλάξετε νοοτροπία. Ευχαριστώ. Thank you. Last speaker. Ευχαριστούμε. Ο Μιχάλη Τιάγκο Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις ε, θέλω να κάνω και μία ερώτηση. Πώς ε, δεν γίνονται αποδεκτά τα προφανή. Λοιπόν, Πρωτο, Πορτογαλία όλοι νομίζω θα συμφωνήσουν. Ήταν ε, ε πειραματόζω. Ε, για τις, ε, τους κοινού κανόνες ε, για την οικοδόμηση της Τραπεζικής Ένωσης και για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τίποτα δεν συνέπεσε όμως με τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας πανήφε με την πτώχευση και την εκαθάριση της τράπεζας αυξήθηκε το δημόσιο χρέος με βάση των επιταγών της, των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ε, η τράπεζα εντάχθηκε στο Σανταντέρ ε, ε, χωρίς να πληρώσει τίποτα. σε μια πολύ μεγαλύτερη τράπεζα δηλαδή ενσωματώθηκε. Και μας λένε ότι αυτό είναι θεωρία συνωμοτική των κομμουνιστών. Ε, τελικά όμως αυτό γίνεται. Συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα, ε, τη μεγαλύτερη. Ε, ε, καθαρίσανε την μικρή τράπεζα και την ενσωμάτωσαν στη μεγαλύτερη. Τι είναι αυτό, δεν είναι συγκέντρωση. Και εμείς τι κάνουμε, απ' την άλλη προσποιούμαστε ότι καταπολεμούμε τους too big to fail και χρησιμοποιούμε την, ε, τελικά την Τραπεζική Ένωση ως εργαλείο ε, ε, και μεθοδεύουμε έτσι την συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι πλέον αριθμισμένος όλων των οικονομικών κλάδων. Και έχει και τα μεγαλύτερα προβλήματα και φέρνει τις μεγαλύτερες ζημιές ε, για όλους, όπως ε, ε, σωστά είπανε όλοι, γιατί το μάρμαρο το πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Αυτά τα ελεπάλληλα στρώματα ρυθμίσεων και μηχανισμών τελικά έχουν ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι, οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών να βρίσκουν παρόλα αυτά παράθυρα και να παρακάμπτουν ε, τη νομοθεσία γιατί δεν είναι βιώσιμα τα συστήματα σε σχέση με το επενδύθεν κεφάλαιο. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να το κράτος να ελέγξει την τράπεζα. Σε αυτό καταλήγουμε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε το αντίθετο, δηλαδή την οικονομία αν θέτουμε στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, Ούγκο Μπάση. Για τις τράπεζες η θα την πάρει ο Ανδρέα. Αλλά έχω να σας πω προσωπικά τα εξής. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά ε, τις ε, απαιτήσει για το reporting που αυτών των εκθέσεων και αναφορών, ε, και εδώ ε, είναι θέμα αναλογικότητα, αλλά θα πρέπει να τα πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα από ό,τι πριν. Ότι θα, φέτος θα γίνει μια σφαιρική, γενική, πλήρης αξιολόγηση των σχετικών απαιτήσεων, ούτω ώστε να, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτήν την πολιτική, όπως την εξήγησε ε, και, και, και, και ρώτησε σχετικά ο κύριο Μπάλτ. Είπαμε ότι θα περιστήλουμε τα προπετούμενα όπου χρειάζεται και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις εποπτικές αρχές. Τώρα έχουμε ξεκινήσει ε, κάποια προτυποποίηση των ε, δεδομένων για να υπάρχει για τα σχετικά δεδομένα, για τα χρηματοοικονομικά δηλαδή, κάποια εναρμόνιση και αυτό αφορά και τους διάβλους της υποβολής των εκθέσεων και αναφορών και έτσι. Αυτό από πλευρά των ρυθμιστικών έργων. Τώρα όσον αφορά αυτά τα ενημερωτικά φυλάδια, τα προσπέκτους, ε, σας υπενθυμίζω ότι είχαμε προτάσεις ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτάσεις ακόμα πιο φιλόδοξες, γιατί θέλαμε ένα κατόφλι ακόμα πιο ε, ψηλό. Και δεν θα ισχύσουν αυτά τα οποία θέλαμε εμείς, ένα ένα, ένα πλήρες προσπέκτους. Έτσι έγινε με την δυναμική της νομοθεσίας, οπότε κατέβηκε ο πύχης των προσδοκιών. Αλλά ήδη με τις δικές μας μελέτες προκύπτει ότι έχουμε ήδη, ήδη μια μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τα προϊσχύσαντα. Και επίσης ε, κλείνω με μια γενικότερη παρατήρηση όσον αφορά την ε, πολυνομία, ε, βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το κατά πόσον πάμε για απορρίθμιση ή ε, αν ήδη έχουμε φτάσει τη, φάση της πολυνομίας αλλά θέλω να σας ε, πω απλώς το ότι στις απαντήσεις για το Call for Evidence γιατί ακούσαμε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και γι' αυτό καταλήξαμε ότι αυτό που προέκυψε όσον αφορά την νομοθεσία είναι ότι τα πράγματα είναι μια χαρά. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο είδου ξεκάθαρη απέτηση, ε, ανάγκη της βιομηχανίας για απορρίθμιση ή για το αντίθετο ή για περισσότερη νομοθεσία. Πάνω κάτω είπαν ότι εντάξει, φυσικά θα πρέπει να πληρώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Άρα πάνω κάτω είμαστε εντάξει. Αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα να κάνει είναι να νομοθετήσουμε όχι περισσότερο αλλά καλύτερα. Μία και δέκα το αργότερο θα πρέπει να κλείσουμε γιατί θα φύγουν οι διερμηνείς. Εν Ευχαριστώ. Πρώτα θα απαντήσω για στην ερώτηση για την εκαθάριση ε, και τη συγκέντρωση διασυνοριακά, δηλαδή για το θέμα του big to fail. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του τραπεζικού τομέα και για την αυτή, αυτοκινητοβιομηχανία και για άλλους ε, ε τομείς που διέρχονται κρίση με πλεόνασμα δυναμικότητας. Ε, το ίδιο σημαίνει. Πρέπει να μειωθεί η δυναμικότητα και η συγκέντρωση είναι μέρος της διαδικασίας. Ε, δηλαδή, το ότι υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση δεν είναι αρνητικό και ότι υπάρχει ενοποίηση διασυνοριακή, ούτε και αυτό είναι αρνητικό. Εφόσον έχουμε ενία αγορά και αυτό είναι σημάδι μεγαλύτερης ολοκλήρωσης, το too big to fail είναι άλλο κεφάλαιο. Φυσικά πρέπει να είναι ισχυρότερε οι δικλείδε ασφαλεία σε αυτή περίπτωση. Αυτό κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν, ε, είναι, αν αυξάνεται το μέγεθο, χρειάζεται ε, περισσότερο κεφάλαιο, χρειάζονται buffers ε, για το συστημικό κίνδυνο, μεγαλύτερο και, και κεφάλαιο, μια υπερδομή που θα μπορεί να καθαρίζεται και εάν ε, ε, συντρέξει ανάγκη, χωρίς να πληρώσουν οι φορολογούμενοι, θα πρέπει να βγαίνετε από την αγορά. Αυτό επιδιώκουμε. Ε, στις μεγάλους συνοριακούς ομίλους δεν έχει δοκιμαστεί το νέο σύστημα, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε και νομίζω είναι θετική εξέλιξη. Επειδή πολλά άκουσα για το δημόσιο χρέος και για το έντες εγγύηση καταθέσεων κτλ. Εάν έχετε ένα ευρώ εγγυήσεων σε μια χώρα που έχουν μικρότερη αξία ή έτσι εκτιμούνται σε σχέση με μια άλλη ευρωχώρα λόγω της ε, ανεπίσημης εγγύησης ε, του κράτους, ποτέ δεν θα έχουμε τραπεζική ένωση. Οπότε χρειάζεται ένα ενοποιημένο σύστημα γιατί αλλιώς ποτέ δεν θα ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση. Γι' αυτό έκανε τις προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το χρονοδιάγραμμα δεν ναι, θα το αποφασίσω εγώ. Υπάρχει το θέμα περιορισμού κινδύνου, των δημοσίου χρέους και εκεί θα πρέπει να κάνουμε κάτι δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος για την φεροεγγυότητα, διότι εφαρμόζονται εσωτερικά μοντέλα για την εγγύηση των δημοσίων ομολόγων. Πολύ διαφορετικές διδαξίες ανάλογα με την τράπεζα, ανάλογα με το κράτος μέλος. Ε, ε, το 11 αρχίσαμε να μιλάμε για την έκθεση για τις ε, κεφαλαιακές ε, απαιτήσει ε, για την έκθεση που σχετίζεται με δημόσιο χρέος και τότε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της κρίσης δημοσίου χρέους και επίσης στην Επιτροπή Βασιλείας και στην Ευρώπη γίνονται κινήσεις για να επιβληθούν απαιτήσει. Αυτό εξυπακούεται όταν υπάρχει κίνδυνος. Εάν χρειαζόμαστε οδικό ε, χάρτη για να δούμε που, ε, ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε, ας το κάνουμε. Ε, για την ε, ρύθμιση. Υπήρχε η ιδέα ότι μπορεί κάποιος να προσελκύσει οι πελάτες αν συρρυκνώσει τις απαιτήσεις, τις ρυθμιστιακές απαιτήσεις για να αντιμετωπίσει το credit crunch. Αλλά Νομίζω ότι ε, φάνηκε ότι αυτό ε, δεν ήταν σωστό. Ε, νομίζω ότι αντλήσανε τα διδάγματα οι μεγάλοι του τομέα που τώρα έχουν αυστηρότερες ε, απαιτήσει γιατί ακριβώς έχουν πολύ μεγαλύτερο ύψος συναλλαγών σε σχέση με το ΑΕΠ, σε σχέση με το, το, το, κεφάλαιό τους. Και έτσι πρέπει να παραμείνει το σύστημα. Ευχαριστούμε, πολύ σύντομα τρία σημεία για τις εγγυήσει επειδή ε, πολλοί είπανε ότι ε, δεν συμβαίνει τελικά σε τίποτα σε αυτό το τομέα παρά τις προσπάθειες. Δεν ισχύει αυτό. Ε, ε τώρα εφαρμόζονται ε, σχεδόν πλήρως οι δύο πρώτοι πυλώνες και όντως πρέπει να καλύψουμε το κοινό και τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει, όχι μόνο πρέπει να τους εφαρμόσουμε, αλλά και να τους χρησιμοποιούμε στην πράξη. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καθυστέρησης ε, στον τομέα της εγγύησης ε, των καθαθέσεων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεύτερο σημείο, ο συνάδελφος από την Πορτογαλία. Μας είπε ότι ήταν η Πορτογαλία για την εφαρμογή των κανόνων. Εγώ αλλά πιστεύω, πιστεύω πως ε, τελικά χρησιμοποιήθηκαν αυστηρότατοι κανόνες ε, που φυσικά για πολλούς ήταν καινούργιοι και στην Πορτογαλία δύσκολα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ε, την ανάγκη τους γιατί ήταν επώδυνοι αυτοί οι κανόνες αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήσασταν και πειραματόζω και εργαστήριο εφαρμογής των νέων ιδεών. Ε, να σταθώ σε αυτό που είπε ο συνάδελφο Κόμπορν. Με το Brexit, λέτε, θα επισπευστεί την κατάσταση επιχειρήσεων. Ε. Ε, ε, υπάρχει αυτή η άποψη, η οποία όμως δεν ξέρω αν ευσταθεί, διότι βλέπουμε ότι υποτίθεται ότι οι διάφοροι θα πρέπει να εκτοπίσουν τις δραστηριότητες τους εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και να τις μεταφέρουν σε άλλα κράτη-μέλη. Θα δούμε όμως ε, τους επόμενους μήνες τι θα γίνει ε, και άλλα παραδείγματα, δηλαδή στο χρηματοπιστωτικό τομέα, μάλλον τελικά το, αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας από το χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι θλιβερό αυτό, αλλά μάλλον αυτή θα είναι η επίπτωση του Brexit. Ε, και ε, είσαστε και συνυπεύθυνοι στο κόμμα σας, ε, κύριε Κόμπορν, για αυτές τις εξελίξεις. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ε, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε Ευχαριστώ τους εθνικούς βουλευτές, ε, τους ευρωβουλευτές. Μπορούμε να πάμε να φάμε και να συνεχίσουμε στις 3 και να συνεχίσουμε με τη διάσκεψη που διεργάζονται με βάση το άρθρο 13. Ευχαριστώ.